ενίσχυση πρέπει ε, να είναι εκ μέρου των λαών μας, των πολιτών μας και όχι μόνο ε, και για τους πολίτες μας και όχι μόνο για τις εταιρείε και αυτό είναι ε, το επίκεντρο της απόφασής μας. Έκλεισε η συζήτηση και το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η εισήγηση Ταραμπέλα, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχετε κύριε Ταραμπέλα για τέσσερα λεπτά το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα ε, να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαίρετη έκθεση. Αυτή η έκθεση που υιοθετούμε κάθε χρόνο έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα. Ε, εγώ είναι η πρώτη έκθεση που παρουσιάζω στην Επιτροπή Γυναικών και είναι απαραίτητη η έκθεση αυτή λόγω της ε, οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ε, τονίζω εδώ τις συνέπειες πάνω στις γυναίκες. Μια διαπίστωση. Οι άνδρες στην αρχή της κρίσης είχαν να υποφέρουν από περισσότερες απολύσεις, αλλά αυτό είναι φυσικό διότι εργάζονται στη βαριά βιομηχανία, αλλά τώρα αυξήθηκε το ποσοστό ανεργίας των γυναικών με τον ίδιο ρυθμό. Σε καμιά δεκαριά κράτη-μέλη το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι ανώτερο και υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες ε, κυρίως στην μερική απασχόληση. Πρέπει λοιπόν να δούμε τις συνέπειες πάνω στους άνδρες και στις γυναίκες και μετά θα πρέπει ε, να γίνουν αναλύσεις αντικτύπου στα κράτη-μέλη ώστε να υπάρχει μια πολιτική ούτω ώστε να μην πλήττονται δυσανάλογα οι γυναίκες. Σε δεύτερο σημείο σημαντικό είναι η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. 20-25% των Ευρωπαίων γυναικών υποφέρουν από βία σωματική ε, στην ζωή τους και 10% σεξουαλική βία θα πρέπει οι άνδρες να δεσμευθούν να ε, προστατεύσουν τις γυναίκες από την βία. Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ε, να δώσει μεγάλη προτεραιότητα σε αυτό το θέμα, δημιουργώντας ένα παρατηρητήριο για την βία κατά των γυναικών, ώστε να υπάρχουν εναρμονισμένοι κανόνες και για να υπάρξει προστασία των θυμάτων. Ζητώ να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, ούτως ώστε όλα τα κράτη-μέλη να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του θέματος αυτού και ο αγώνας αυτός να γίνει μια προτεραιότητα. Απασχόληση, 59,1% ε, των γυναικών εργάζονται σήμερα ε, είχαμε στην στρατηγική της Λισαβόνας ένα στόχο 60%, τον πλησιάζουμε, αλλά υπάρχει διαφορά ανάλογα με τα κράτη-μέλη και επίσης διαφορά στις αμοιβέ που σύμφωνα με τις μελέτες είναι από 17-25%. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουν τις οδηγίες ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της απασχόλησης και να λάβουν μέτρα νομοθετικά για να ευνοήσουν μια ισορροπημένη παρουσία των ανδρών και γυναικών στις θέσεις ευθύνη επιχειρήσεις, κυρίως στις ε, ιδιωτικές εταιρείες. Σχετικά με τις συμπεριφορές τις σεξιστικές, εγώ ως υπουργό Πληροφοριών, μια γυναίκα έπρεπε ε, να σταματήσει την ε, ε, εκπαίδευσή της ως οδηγός λεωφορείου σχολικού λόγω του γεγονότος αυτού. Κανείς δεν θα πρέπει να εκπλήσεται τώρα ένας άντρας να πλένει τα πιάτα ή μια γυναίκα να οδηγεί ένα σχολικό λεωφορείο. Πρέπει να υπάρξουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης στα σχολεία προς το θέμα αυτό. Σεξουαλικά δικαιώματα και αναπαραγωγής θα πρέπει οι γυναίκες να μπορούν να ελέγχουν ελέγχουν ε, το, το, το, την κατάσταση αυτή. Πάρα πολλέ γυναίκε αγωνίστηκαν με κίνδυνο τη ζωή του. 24 χώρε, 27 έχουν τώρα νομιμοποιήσει ε, τι αμβλώσει ε, και θα πρέπει να βοηθήσουμε τις ε, γυναίκες ε, και οι γυναίκες θα πρέπει να ελέγχουν τα δικαιώματα αυτά, να έχουν πλήρη δικαιώματα προς τη σεξουαλική του ζωή και την αναπαραγωγή και τις αμβλώσεις. Η, ε, η άδεια στους, στους πατέρες για, την λογοτεκνοποίηση θα υπάρχει λοιπόν μια ευρωπαϊκή άδεια και θα πρέπει ε, σε περίπτωση τεκνοποίησης της γυναίκας να μπορεί και ο πατέρας να πάρει άδεια. Η έκθεση αυτή επενέθηκε από πάρα πολλούς, από ε, πολλές ομάδες πολιτικές στην Επιτροπή Γυναικών. Υιοθετήθηκε η έκθεση αυτή με μεγάλη πλειοψηφία. Καλό λοιπόν όλους τους συναδέλφους να υποστηρίξουν στην ψηφοφορία την Τετάρτη την έκθεση αυτή, αλλά ε, παρόλα αυτά θα παρακολουθήσω με πάρα πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση και θα μπορούσα να απαντήσω στην συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Ταραμπέλα. Ο κύριος Σπίτλα έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές. Η Κομισιόν αποδέχεται την έκθεση για την ισότητα για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη το 2009 ε, ευχαριστώ για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έκθεση της Κομισιόν. Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απαράβατο όρο για την υλοποίηση των στόχων της κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης στην Ένωση. Σε αυτή τη βάση η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδόμησε μια πραγματική πολιτική ισότητας μεταξύ των φύλων. Αν, αν και αδιαμφισβήτητη η πρόοδο στον τομέα αυτό, οι προκλήσεις είναι τεράστιες και συμμερίζεται η Κομισιόν τη γνώμη του εισηγητή. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες κατά την δική μου θητεία η ισότητα των φίλων ήταν το θέμα που είχα πραγματικά στην καρδιά μου και την τελευταία πενταετία είχαμε συγκεκριμένη παρέμβαση με την roadmap για την ισότητα και την προσπάθεια υλοποίησης αυτών των μέτρων πάλεψε η Κομισιόν για να μειώσει τη διαφορά των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών που είναι 17% και είναι απαράδεκτο. Στο μέλλον η Κομισιόν θα παρουσιάσει προτάσεις για την εξάλληψη των ανισοτήτων στους μισθούς και θα βάλει ως παράδειγμα το ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Τον Μάρτιο του 2009 η Κομισιόν θέλησε να κινητοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους για τον ίσο μισθό και επειδή αυτή η εκστρατεία έχει ιδιαίτερη επιτυχία θα συνεχιστεί και το 2010 θέλουμε επίσης να έχουμε μεγαλύτερη προσώπηση των γυναικών στον οικονομικό και πολιτικό βίο και τον Ιούνιο του 2008 δημιούργησα ένα δίκτυο γυναικών leader. Pourtant 35% των γυναικών αντιπροσωπεύονται στην πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά στις χώρες είναι το ποσοστό αυτό κάτω του 25% και μόνο το 11% είναι στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων ε, των μεγάλων επιχειρήσεων που βρίσκονται στο χρηματιστήριο. Χρειάζεται λοιπόν ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και χαίρομαι σήμερα όμως που λέω ότι το σχετικό Ιστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων ξεκίνησε τις εργασίες του στις Βρυξέλλες και έχει εγκατασταθεί στην Αβενή Λουίζ. Λοιπόν, πρέπει μέσα στο γενικό πλαίσιο της ε, κρίσης να προστατεύσουμε τη γυναικεία απασχόληση. Επίσης θα πρέπει να συνδυάσουμε την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή και συμφωνώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που υπογραμμίζει τον ρόλο του πατέρα που θα πρέπει να αναβαθμιστεί μέσα στην οικογένεια και γι' αυτό ζήτησα από τις υπηρεσίες μου να κάνουν μία μελέτη για το κόστος ωφέλεια μίας παρέμβασης της Κομισιόν στον τομέα αυτό. Επίσης, πρέπει να σταματήσει η βία κατά των γυναικών. Η Κομισιόν λοιπόν θα εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση με σθένος και παλμό. Δεν θέλω να σταματήσω την τοποθέτησή μου χωρίς να αναφέρω την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν που αποτέλεσε ουσιαστικότατο παράγοντα για την πρώτη θέση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν είναι αυτός σκοπός πρέπει να συνοδεύεται από απασχόληση και κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας. Ευχαριστώ Επίτροπε. Ξεκινάμε λοιπόν με το ΕΛΚ, δύο λεπτά την κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Πρόεδρε, με έξι απόντες, απούσες τους 33, ε, υπερψήφισε η έκθεση, την έκθεση αυτή. Εμείς συμμεριζόμαστε όλες αυτές τις ανησυχίες για τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και αυτό παρά το ότι έχουμε μια πολύ καλή νομοθεσία, κοινοτική νομοθεσία από το 1975 και μετά στον τομέα αυτό. Γιατί λοιπόν διακρίσεις που μας κάνουν τη ζωή δύσκολη, είτε γιατί οι οδηγίες εφαρμόζονται άσχημα, είτε γιατί αυτές που υπόκεινται τις διακρίσεις δεν πάνε στα δικαστήρια. Έτσι λοιπόν εμείς τι γίνεται. εκπονούμε οδηγίες και άλλες οδηγίες και μπερδεύουμε ακόμη περισσότερο το εθνικό νομικό πλαίσιο χωρίς να πετούμε ήδη υπάρχουσες οδηγίες να εφαρμόζονται σωστά και από τα κράτη-μέλη και από τους κοινωνικούς εταίρους και στον καθημερινό βίο. Και κάθε μέρα άντε γενικολογίες για τις γυναίκες που τρών ξύλο, που τις βιάζουν, που καταπιέζονται στην οικογένεια και άντε πάλι εκθέσεις και κόντρα εκθέσεις και τροπολογίες και κόντρα τροπολογίες και Όλοι θεωρούν ότι άμα βρουν οι γυναίκες δουλειά και απασχόληση τότε θα έχουμε και την πανάκια ότι οι γυναίκες θα ανεξαρτητοποιηθούν μέσα από την οικονομική απολευθέρωση η τώρα Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Τι θα γίνει, θα δημιουργήσει νέα γραφειοκρατία. Λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία είναι ασύμβατη με την ισότητα των φίλων που έχει μπει και στη συνθήκη. Αν πραγματικά το γελίο δολοφονεί ε, πραγματικά βρισκόμαστε σε τέτοιου είδους παράδειγμα λέει Δηλαδή και αν θεωρείτε εσείς ότι η αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία συμβαδίζει με τις εκτρώσεις, ε όχι βέβαια, γελιέστε. Θα πρέπει να μιλήσετε περισσότερο για την αντισύλληψη που στον καιρό μου δεν υπήρχε. Και η αντισύλληψη είναι αυτή που θα μας οδηγήσει στην αποφυγή ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών που στον καιρό μου δεν υπήρχε. Αλλά ο κύριος Ταραμπέλα εδώ έπεσε θύμα του εξτρεμισμού των συντρόφων του, έστω και αν δεν είναι γυναίκα ο ίδιος. Ευχαριστώ. Για τους σοσιαλδημοκράτες η κυρία Γκαρσία Πέρες για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον κύριο Ταραμπέλα για την έκθεσή του και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην επεξεργασία αυτής της έκθεσης. Πριν από ένα χρόνο εμείς συζητούσαμε μία αντίστοιχη έκθεση με αυτή που έχουμε μπροστά μας και δυστυχώς θα πρέπει να συνεχίσουμε να επιμένουμε γύρω από ουσιαστικά θέματα τα οποία δεν καταφέραμε σε ένα χρόνο να προχωρήσουμε για θέματα ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών η ανισότητα αποτελεί μάστιγα όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον κόσμο. Αυτή η διαφορά μισθών που παραμένει σταθερή και δεν καταφέρνουμε να μειώσουμε. Τα δικαιώματα στην αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία. Ο συνδυασμός οικογένειας και επαγγέλματος. Η ισότητα στην πρόσβαση στην αγορά οι γυναίκες ε, στην Ήπεθρο, οι γυναίκες ε, με αναπηρία, η παρουσία των γυναικών στο δημόσιο βίο είναι πράγματα που τα λέμε και τα ξαναλέμε κάθε χρόνο και δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε. Ένα στοιχείο να σας αναφέρω. Μόνο τρει από τα 27 κράτη-μέλη έχουν πάνω από 40% γυναίκες βουλευτές στα κοινοβουλίο τους. Λοιπόν, θα πρέπει να επιμείνουμε ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι ουσιαστικό να προχωρήσουμε σε πρωτοβουλίες σαν αυτή της Ισπανικής Προεδρίας που έχει ως προτεραιότητα την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πρόκειται για μια στράτευση όχι μόνο δική μας αλλά και για τις μελλοντικέ γενιές. Ήδη κάναμε μια μεγάλη πορεία. Θα πρέπει όμως να παλέψουμε ούτως ώστε το μισό του πληθυσμού της Ευρώπης να έχει τέλεια δικαιώματα με το υπόλοιπο μισό. Για τους φιλελεύθερους η κυρία Ιντβελτ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή. Τούτου λεχθένω όμω θα ήθελα να αναφέρω και κάποια σημεία με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί σα όσον αφορά τι επιπτώσει παραδείγματο χάρη τη οικονομική κρίση στι γυναίκε. Θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ξυγιάνουμε τα δημόσια οικονομικά γιατί αυτό είναι προ όφελο των γυναικών. Όχι να αυξήσουμε το δημόσιο χρέο, αυτό δεν οφείλει κανέναν. Υπάρχουν επίση κάποιε προτάσει στην έκθεση που έχουν κάπω ένα συμβολικό χαρακτήρα ένα έτος υπέρ του ενός και του άλλου ή κέντρα επιτήρησης για τούτο και το άλλο. Εγώ θέλω να έχουμε πολύ συγκεκριμένα θέματα. Θα σας πω τι μου αρέσει πολύ. Καταρχήν, χάρη σε μια τροπολογία της Άλτερ, έχουμε μία αναφορά στις μονογονικές οικογένειες και θα ήθελα να κάνω εδώ μία έκκληση προς την Κομισιόν να κάνει μία σχετική έρευνα γιατί έχουμε μία ευρωπαϊκή πολιτική οικογένειας κανένας όμως σχεδόν δεν γνωρίζει ότι κάθε τρίτο νοικοκυριό στην Ευρώπη είναι μονογονικό. Πού πλήττεται όσον αφορά τα φορολογικά θέματα, την κοινωνική ασφάλεια, την κατασκευή οικίας κλπ. Τρίτον, εγώ και στρέφομαι στην κυρία Λούλη, χαίρομαι ιδιαίτερα που αναφέρεται εδώ η σεξιολογική και μου στην κυρια λουλη χαιρομαι ιδιαιτερα που αναφερεται εδω η σεξουαλική και αναπαραγωγικη ε, ανεξαρτησια της γυναίκας και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει πρόσβαση και σε σίγουρη και νόμιμη άμβλωση. Ε, συμφωνώ με την κυρία Λούλη. Είναι σημαντικό να ε, είναι κανένας καλά ενήμερο, αλλά στη χώρα μου, δεν ξέρω τι γίνεται στο Λουξεμβούργο, στη χώρα μου τουλάχιστον αυτό υποσκάπτεται από τους φιλοδημοκράτε. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε μαζί για να ενημερώσουμε καλύτερα τι νέε γυναίκε και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ξέρετε ότι θα έχετε την υποστήριξή μου. Θα πρέπει να ε, μην ε, τιμωρούμε τις γυναίκες ή να τις ε, ε, υποχρεώνουμε να έχουν πολύ επικίνδυνες απλώς γιατί μυστικές κλπ. Τέλος θα ήθελα να σας πω ότι θα χαιρόμουν εάν η Προεδρία του Συμβουλίου βασιζόμενη στην αυτή οδηγεί το σε μία πρωτοβουλία γιατί πολλοί δεν ξέρουν ότι υπάρχει τόσο πολύ βία κατά των γυναικών. Ευχαριστώ για τους πράσινους. Ο κύριος Κορνελίσεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε σχετικά νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχεδόν και μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι Πρώτη φορά με την έκθεση Ταραμπέλα που ψηφίζουμε για το ποια δράση θέλουμε να αναλάβει το κοινοβούλιο αυτό τα επόμενα χρόνια. Η πράσινη είναι πολύ ικανοποιημένη με την αρκετά προοδευτική αυτή η έκθεση. Ε, συμπεριλαμβάνει μια σειρά σχεδίων που θέλουμε να πραγματοποιηθούν. Τελικά θέλουμε να η νομοθετική δράση για να κατανεμηθεί η φροντίδα των παιδιών ε, και στους δύο γονείς με την πρόθεση της άδειας πατρότητας. Επίσης θα μπορούσαμε να ε, κοιτάξουμε ποια είναι η πρακτική στην Ορβηγία όσον αφορά τις ποσοστώσεις η, ε, ανάμεσα στα δύο φύλλα για πολλές ε, από τις οδηγίες. Επίσης θα πρέπει να δούμε τις επιπτώσεις της κρίσης στις γυναίκες. Ε, τα ποσοστά ανεργίας είναι διαφορετικά από εκείνα των ανδρών και οι επιπτώσει περικοπής των ε, δημοσίων δαπανών στις γυναίκε επίση διαφέρουν από κοινέ στου άντρε. Ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο θα δειχθεί τολμηρό και πανέτοιμο για να καταπολεμήσει τις διακρίσεις στις βάρος των γυναικών και ίσως να υποβάλει και κάποια σχέδια που θα οδηγήσουν σε αποτέλεσμα. Θα υπερψηφίσουμε την έκθεση αυτή και ελπίζω πραγματικά η Κομισιόν να αναλάβει τη σχετική δράση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τους συντηρητικού, ο κύριο Σιμάνσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι με την έκθεση αυτή γίνεται πιο ε, ε, διαδίδεται, διαδίδονται οι αμβλώσεις και μειώνονται τα δικαιώματα των χωρών να ασχοληθούν με αυτόν τον τομέα. Δεν χρειάζεται κανείς να προχωρήσει πολύ ε, και μπορεί κανείς ακόμα στο πιο μικρή βελγική πόλη ε, να δει πόσο συχνές είναι αυτές οι υπορριπτώσεις ε, με τους υπέρηχους ε, και θα πρέπει οι υπεύθυνε αρχές να κάνουν ό,τι μπορούν για να μειωθεί ο αριθμός των αμβλώσεων. νομίζω ότι παρεκκλίνουμε από τον ανθρωπισμό επιτρέποντας τόσες πολλές αμβλώσεις. Ευχαριστώ για την ΓΟΕ. Η κυρία Φιγκερέιδο για μισή λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως αποδεικνύει η πραγματικότητα και το επιχειρώνει και η η οικονομική κρίση πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες, αυξάνεται η ανεργία, αυξάνονται οι κακοπληρωμένες και προσωρινές δουλειές, αυξάνεται το χάσμα του μισθού μεταξύ ανδρών και γυναικών, ξεπερνάει και το 17% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει φτώχεια λόγω των χαμηλών μισθών και εισοδημάτων. Η μεταρρύθμιση των συντάξεων επίσης δεν είναι υπέρ των ε, γυναικών οι οποίες με δυσκολία μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες. Μετά έχουμε την πορνεία, τη σωματεμπορία, την οικογενειακή βία, την διάκριση των γυναικών σε όλους τους τομείς. Όπως λέγεται στην έκθεση και συγχαίρω τον εισηγητή γι' αυτό, είναι σημαντικό να προσέξουμε <coughs> την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των γυναικών όταν επεξεργαζόμαστε κοινωνικές ε, και οικονομικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως όταν πρέπει να μελετήσουμε τις κοινωνικές επιπτώσεις για να εγγυθούμε η ισότητα και κοινωνική πρόοδο και όχι οπισθοχώρηση. Πρέπει να προστατεύσουμε την μητρότητα και την πατρότητα πρέπει να στοιχηματίσουμε σε μια στρατηγική ανάπτυξης και κοινωνικής πρόοδου που θα δίνει προτεραιότητα σε δημόσιες υπηρεσίες ποιότητας και κοινωνική ενσωμάτωση. Πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα μπρος για να προστατεύσουμε τις γυναίκες και για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία σταματώντας με τις υποκρισίες που υπάρχουν ακόμα σήμερα για τα θέματα των αμβλώσεων για την Ευρώπη ελευθε, της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας ο κύριος Μπάτεν για 1,5 λεπτό. Υπάρχει μια ιδεολογία που κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη που ε, διδάσκει την ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, λέγοντας ότι οι γυναίκες είναι κατωτέρου επίπεδου από τους άνδρες, ότι ε, θα πρέπει λοιπόν να έχει διπλή μερίδα ο άνδρας από τις γυναίκες λένε ότι ε, σε ένα δικαστήριο η μαρτυρία δύο γυναικών ισούται προς τη μαρτυρία ένα, ενός, άνδρας, ενός άνδρα. Αλλά η, ε, και πως πολλές φορές η μαρτυρία μιας γυναίκας ε, δεν γίνεται δεκτή. Ε, και στον Ισλαμικό κόσμο οι τέσσερις άνδρες των οποίων η μαρτυρία έχει σημασία ε, είναι ε, άνδρες. Αυτός είναι ο νόμος της Σαρία όπου η μαρτυρία μιας γυναίκας δεν έχει, δεν έχει καμία χρησιμότητα. Βεβαίως, εκεί είναι κατάφορη περίπτωση παραβίασης της ισότητας μεταξύ των φίλων η Βρετανική κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει την ομοθετησάρια Σάρια σε ορισμένα δικαστήρια και ενώ η διγαμία είναι νόμιμη ε, στην ε, Μεγάλη Βρετανία ε, και γίνεται πολύ συχνά για απαλλαγές φορολογικές. Εάν θέλουμε πραγματική ισότητα, θα πρέπει τα μεμονωμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην αναγορίζουν τον νόμο της ε, Σαρία, κατ' ουδένα τρόπο. Ευχαριστώ για τους μη εγγεγραμμένους. Ο κύριος Βέρτμαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. περισσότερες γυναίκες είναι στην αγορά απασχόλησης, όμως ε, μια αύξηση το θέση να απασχολήσει σημαίνει να αυξάνει και η ποιότητα των να απασχόληση. Πολλέ γυναίκε εργάζονται σε μερική απασχόληση ή σε εργασίε οι οποίε πλήττονται ιδιαίτερα από τη σημερινή κρίση. Περίπου το 60% εκείνων που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια είναι γυναίκε, αλλά υπάρχουν εμπόδια για τι γυναίκε που δεν του επιτρέπουν να εκμεταλλευτούν τι δυνατότητέ του πλήρω. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχουν ορισμένα δεσμευτικά ελάχιστα πρότυπα ελάχιστες ε, προδιαγραφές για την άδεια μετά τη γέννηση ενός παιδιού, βελτίωση της ε, φροντίδας στο σπίτι κλπ. Έτσι μπορούν να καταρριφθούν κάποια, ε, κάποιες συνήθειες και να προχωρήσουμε πολύ πλησιέστερα στην ισότητα άνδρων και γυναικών. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε στο κατάλογο των άλλων γεγραμμένων ομιλητών. Θα αρχίσω κυρία Μπάουερ για δύο λεπτά. Είμαι βέβαιη ότι ο κύριος Ταραμπέλα θα με συγχωρήσει αν δεν του πω ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα πω ευχαριστώ στον κύριο Σπίτλα, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ μας για τελευταία φορά ως Επίτροπος. Επιτρέψατε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο για τη δέσμευσή του. Ήταν πάντοτε δεσμευμένος, στρατευμένος για τις γυναίκες, για το ρόλο των γυναικών στην αγορά εργασίας και υπέρ της ισότητας των ευκαιριών για τις γυναίκες. Και σχέση με το κείμενο θα ήθελα να αφερθώ σε δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα η διαφορά μισθών ανάμεσα στους άνδρους και στις γυναίκες. Είναι πάνω από 17 7% η διαφορά. Η κατάσταση αν βελτιώνεται, βελτιώνεται βραδύτατα και πρέπει να σας πω ότι τα στοιχεία είναι χειρότερα από ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια. Αν κοιτάξουμε την κατάσταση την καθημερινή, νομίζω ότι βραχυπρόθεσμα δεν μπορούμε να περιμένουμε καμία βελτίωση. Και αυτό που είναι τελείως απαράδεκτο είναι ότι η διαφορά δεν παρουσιάζεται στους νέους, αλλά παρουσιάζεται πολύ περισσότερο για τις γυναίκες που προσπαθούν να επανανταχθούν στην αγορά εργασίας αφού έχουν τεκνοποίηση. Σε αυτή την Ευρώπη, η οποία έχει πληγεί από την κρίση, είναι απαράδεκτο αυτό. Βεβαίως, η διαφορά αυτή απαγορεύεται από πάρα πολλούς κανόνες και επίσης ε, μιλήσατε για την ε, νομοθεσία του 75 και για την οδηγία η οποία υπάρχει εδώ και καιρό, αλλά αυτή η οδηγία παρόλο που υπάρχει δεν είναι αποτελεσματική. Χάρηκα που ο κύριος Σπίτλα είπε ότι μπορούμε να περιμένουμε μια σημαντική έκθεση από την Επιτροπή για το 2010. Σε αυτήν την έκθεση η Επιτροπή θα μας εξηγήσει τι προτίθεται να κάνει ούτως ώστε η νομοθεσία να γίνει πιο αποτελεσματική. Και επιτρέψατε μου να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με τον χάρτη των γυναικών, με την ισότητα των γυναικών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης νομοθεσίας. Αυτό είναι καλύτερο από το να δημιουργούμε νέες νομοθεσίες που θα είναι εξίσου αναποτελεσματικές όπως οι παλαιότερες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Στρέλα, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική του εργασία και ελπίζω ότι οι προτάσεις που θα προκύψουν από αυτό το ψήφισμα θα εγκριθούν. Κατά το ευρωπαϊκό έτος ε, για την καταπολέμηση της στόχης και τον κοινωνικό αποκλεισμό διαπιστώσαμε ότι το πρόσωπο της φτώχειας είναι περισσότερο, όλο ένα και περισσότερο γυναικείο. Οι περισσότεροι φτωχοί στην Ευρώπη είναι γυναίκες και παιδιά. Με την οικονομική και κοινωνική κρίση είναι η κατηγορία που υποφέρει περισσότερο από όλου. Οι γυναίκες είναι οι τελευταίε που μπαίνουν στην αγορά εργασία και είναι οι πρώτες που παίρνουν δρόμο για την ανεργία. Πρέπει επίσης να προσθέσουμε ότι το 2004 μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν του 15% και το 2009 πάνω από 17%. Θέλω να επιστήσω λοιπόν την προσοχή σας και να ζητήσω την υποστήριξη των συναδέλφων για ορισμένες προτάσεις που θεωρώ ότι αποτελούν καινοτομία και είναι και σημαντικές. Πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή χάρτα των δικαιωμάτων των γυναικών που λείπει. Ε, Μία πρόταση οδηγίας ε, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, δηλαδή σωματεμπορία και οικογενειακή βία στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα πρέπει να μπει και η άδεια πατρότητας όχι μόνο μητρότητας όπως ισχύει και σε πολλές χώρες για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε καλύτερα την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή όπως επίσης και να προωθήσουμε την τις ε, γεννήσεις. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Επίτροπο Σπίτλερ για όλη τη συνεργασία αυτά τα χρόνια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Παρμάνοβα για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή. Είμαι πεσμένη ότι αυτή η έκθεση δίνει τη σωστή απάντηση σε διαφόρων τύπων διακρίσεις κατά των γυναικών. Και αυτό για μένα είναι μια νέα και αποτελεσματική δέσμευση για να εξασφαλίσουμε την ισότητα μεταξύ των φούλων στην Ευρώπη, να προωθήσουμε κοινωνικονομική θέση των γυναικών, ιδίως στα νέα κρατμέλη. Χρειάζεται να υπόψη μας ότι τα θεσμικά όργανα είναι εκείνα που αποφασίζουν στην πρόσβαση των ανδρών ή των γυναικών στους πόρους. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποδείξουμε ότι οι γυναίκες είναι εκείνες που θα μπορούν να παίρνουν τις αποφάσεις στην πολιτική και στις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να εκμεταλλεύονται στα συμβόλια των διευθυντών και θα πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για την εξέλιξη της, νοοτρο... της ε, τους όπως και οι γυναίκες ε, και οι άνδρες Ιδίως μετά από την άδεια μητρότητας χρειαζόμαστε τους ε, θεσμικούς μηχανισμούς που θα κινητοποιήσουν μια συνεπή πολιτική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Γιατί η διάκριση των φύλων μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, στρατηγικά μέτρα και συνέπεια. Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε την ανεργία, ιδίως την ανεργία τύπου Β και να υπάρχει ισότητα για την πρόσβαση σε όλους τους πόρους. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και η Κομισιόν, πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη και την κοινωνία των πολιτών να υιοθετήσουν αποτελεσματικά μέτρα. Είμαι πεπισμένη ότι οι γυναίκες είναι σε θέση να είναι αποτελεσματικές όσον αφορά και τις πολιτικές ε, και τις οικονομικές πτυχές των προβλημάτων και θα μπορέσουν να προωθήσουν την ανάπτυξη στις χώρες τους και την καλή διακυβέρνηση. Με αυτά τα λόγια η προώθηση της ισότητας των φύλων είναι η σωστή λύση για να ξεπεράσουμε την οικονομική και κοινωνική κρίση και να αντιμετωπίσουμε την δημογραφική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Μπραντνερ για ένα λεπτό. Θα ήθελα να τονίσω δύο απόψεις της έκθεσης που είναι σημαντικές για την ομάδα μας. Και ελπίζω τα σχόλια αυτά να τα διαβιβάστε στο νέο επίτροπο. Δύο σημεία. Το πρώτο είναι η αναθεώρηση που έχει ζητηθεί εδώ και πολύ χρόνο της οδηγίας για ίση αμοιβή, για ίση εργασία. Αυτό είναι κρίσιμο για όλες τις γυναίκες σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η διαφορά, η απόκληση είναι σημαντική, είναι απαράδεκτη. Το δίγνυμα βρισκόμαστε στο 2010 πρέπει να γεφυρωθεί αυτή η διαφορά και χρειάζεται νομική δράση. Περιμένουμε προτάσεις της Κομισιό για το μέτρο που θα ληφθεί για να εξασφαλιστεί αυτό. Ε, περιμένουμε ότι θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια αυτής της ε, θητεία. Ε, τώρα όσον αφορά την άδεια θα ήθελα να τονίσω ότι είναι σημαντικό για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Χρειάζεται ισότητα και για τους άνδρες, ε, ότι μπορούν να έχουν χρόνο με, για τα παιδιά τους, ότι να έχουν την ευθύνη αν το επιθυμούν. Χρειαζόμαστε ίση επιλογή για τους άνδρες και για τις γυναίκες για το πώς θα ζήσουν, θα εργαστούν και πώς θα φροντίσουν για την οικογένειά τους και τα παιδιά τους. Πιστεύουμε ότι είναι κρίσιμο ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλει ένα σήμα, ένα μήνυμα στους πατέρες, αλλά θα θέλαμε να στείλουμε περισσότερο από ε, σήματα, να ανοίξουμε τις πόρτες για την σύγχρονη κοινωνία και εξαρτώμεθα από την Κομισιόν για να εισαγάγει ε, μια οδηγία η οποία να είναι σύγχρονη και ανοιχτή περιμένουμε τις προτάσεις της Ισπανικής Προεδρίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στην Ευρώπη και ελπίζουμε η Επιτροπή να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκέρλινγκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Εμείς οι ε, γυναίκες ευρωβουλευτές είμαστε σε μειονότητα ε, έχουμε ικανοποιητική εργασία, ίσες αμοιβέ, ε, ίσα δικαιώματα στα εξωτερικά. Πολύ διαφορετική θέση δηλαδή από ό,τι πολλοί από τις εκλογέ μας. Χαιρετίζω την έκθεση αυτή και χαιρετίζω τις προσπάθειες του κ. Ταραμπέλα και το ότι τονίζει την οικονομική ευημερία των γυναικών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για την ισότητα των φίλων. Οι γυναίκες μπορούν να ελέγχουν οικονομικά τη ζωή τους, θα μπορούν πολύ καλά να ε, ελέγξουν και όλε τι άλλε πτυχέ τη ζωή τους. Θα πρέπει να φροντίσουμε σε αυτούς του τόσο προκλητικούς οικονομικούς καιρού να μην μείνουν πίσω οι γυναίκες με χαμηλή ε, πληρωμή σε ε, πολύ επισφαλείς θέσει απασχόλησης. Θα ήθελα να χαιρετήσω την πρόσκληση που έγινε να σπουδάζουν περισσότερο οι γυναίκες ε, ε, θετικές επιστήμες και να εργαστούν στον τομέα της μηχανικής επίσης. Οι ανάγκες της γυναίκας είναι όσον αφορά τις δράσεις. Η δράση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και οικονομικά θα μπορούν να ορθοποδήσουν. Ευχαριστώ. Κυρία Σμένσον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κύριο Ταραμπέλα και τους συναδέλφους της Επιτροπής για αυτή την εξαιρετική έκθεση. Να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Ελπίζω ότι θα υπάρξει υποστήριξη στο σχέδιο για την άδεια πατρότητας. Η άδεια πατρότητας δεν αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα μόνο για τις ίσες ευθύνε των δυο γονιών, αλλά θα έχει και άλλες θετικές επιπτώσεις όλοι όλα αποδεικνύουν ότι οι πατεράδες οι οποίοι έχουν πάρει άδεια πατρότητας έχουν διαμορφώσει καλύτερες σχέσεις με τα παιδιά τους. Επίσης, οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν οι ίδιες για το κορμί τους, για τη σεξουαλικότητά τους και την αναπαραγωγή τους. Τα παιδιά πρέπει να είναι πρόσδεκτα, να τα θέλει κανείς. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε παιδιού να είναι επιθυμητό. Πρέπει να σταματήσει σήμερα, το φαινόμενο σήμερα γυναίκες να πεθαίνουν στο, στο, στο, στο, στο βωμό των αμβλώσεων. Δώστε δυνατότητα στις γυναίκες να αποφασίζουν όχι μόνο στην οικονομία και στην πολιτική αλλά και για το κορμί τους. Σμιτ για δύο λεπτά. Σημερίζομαι. Σημερίζομαι αυτή τη θέση λοιπόν. Αλλά αναρωτιέμαι γιατί οι γυναίκες πιστεύουν σήμερα ότι ο αγώνας για την ισότητα είναι ένας αγώνας στον οποίο συμμετέχουν μόνο οι γυναίκες. Εγώ χαίρομαι όμως που η ομάδα μου έβαλε δύο άντρες να προστατεύσουν τις γυναίκες και την πολιτική τους. Σήμερα η ισότητα βλέπουμε να αντιμετωπίζεται μόνο στο κοινωνικό και οικονομικό τομέα. Μιλάμε για ίση αμοιβή και ίση δουλειά, αλλά είναι σημαντικό αυτό, αλλά υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι το τεράστιο πολιτιστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην ισότητα και αυτό λόγω της μετανάστευσης από τις Ισλαμικές χώρες. Μιλάμε εμεί σήμερα για ισότητα, αλλά δεν μιλάμε ούτε γίνεται καν νήξη για τους καταναγκαστικούς γάμους, ε, για την κοπή της κλιτορίδας. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να αναφέρονται και να μπαίνουν μέσα στο πλαίσιο της Ευρώπης του 2010 και της κατάστασης των γυναικών. Η κυρία Μόρβαη για ένα λεπτό. Όσον αφορά... Θα ήθελα να σας πω ότι ε, εδώ προτείνουμε μία νέα αντιμετώπιση θα πρέπει πραγματικά να φροντίσουμε να προσφέρουμε καλές υπηρεσίες στις γυναίκες. Οι γυναίκες ξέρουν πολλά. Και εμείς ξέρουμε πολλά για την κατάσταση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ συγκεκριμένα στο θέμα των αμβλώσεων. Οι αμβλώσεις αυτές τις αυτές είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κεφάλαιο για τις γυναίκες και θα ήταν καλύτερα να προλαμβάνουμε, να μην χρειαστεί να φτάνουν στην ε, άβλωση. Πρόληψη λοιπόν είναι η σημαντική, η αντισύλληψη είναι σημαντική. Ε, η εμπλώτηση είναι ε, αποτέλεσμα μιας μία επιθυμητής ε, εγκυμοσύνης και θα πρέπει λοιπόν καλύτερα να εξηγήσουμε στις νέες γυναίκες πώς θα αποφύγουν την εγκυμοσύνη και όχι να προσπαθούμε μετά να τους επιτρέψουμε τις αμβλώσεις. Ευχαριστώ η κυρία Ζαμπόρσκα για δύο λεπτά. Κυρία, κυρία Πρόεδρε, το σχέδιο ψηφίσματος συναδέλφου Ταραμπέλα που ήρθε στην Επιτροπή Γυναικών από τις τελευταίες ευρωεκλογές είναι φιλόδοξο και αναφέρομαι κυρίως στην παράγραφο 20. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί να υπάρξει μια Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα Δικαιώματα των Γυναικών. Αν γνωρίζουμε την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η Συνθήκη της Ρώμης ήδη προέβλεπε το κείμενο του νόμου με την αρχή της ισότητας ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες στην αγορά εργασίας ο νόμος για την ίση μεταχείριση των ανδρών και γυναικών. Ο νόμος αυτός υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη. Μια λύση απλότητας θα ήταν να ζητήσουμε μια νέα χάρτα. Θα μπορούσαμε όμως να εφαρμόσουμε και τα υφιστάμενα μέσα στην πραγματικότητα αν δεν αφαιρέσουμε την παράγραφο 20 από αυτό το σχέδιο ψηφίσματος, τότε προσθέτουμε στην Ευρωπαϊκή Σύμβοση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ε, Συμβουλίου της Ευρώπης την Χάρτα των ε, Δικαιωμάτων και έχουμε ένα τέταρτο μέσο το οποίο εμφανίζεται με την μορφή μιας νέας ιδιαίτερης χάρτας για την πρόθεση της γυναίκας. Έχω μερικές ερωτήσεις. Τι ποια θα ήταν η χρησιμότητα μιας νέας χάρτας των δικαιωμάτων της γυναίκας, ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία της. Δεν υπάρχει καμία. Θα ήταν σφάλμα να πιστεύουμε ότι μια χάρτα θα επιλύσει τα προβλήματα των γυναικών. Το φυσικό δίκαιο που θα πρέπει να υπαγορεύει τον προβληματισμό μας και την υπεύθυνη δράση μας στην πολιτική δεν αναφέρεται σε ιδιαίτερα δικαιώματα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι τα νομικά μέσα αγνοούν τα δικαιώματα της γυναίκες. Θα ήταν ανέντιμο διανοητικά και εσφαλμένο στην πραγματικότητα. Γι' αυτό ψηφίζω κατά της παραγράφου 20 το θέμα της χάρτας Εάν σε αυτό το σχέδιο ψηφίσματος παραμείνει η παραγραφος 20, δεν θα μπορέσω να υποστηρίξω το σχέδιο αυτό. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας με την Επιτροπή των Γυναικών κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκυγιόμ για 1,5 λεπτό. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Μάρκα Ταραμπέλα για την έκθεση και την επιτυχία με την οποία εξετέλεσε την εργασία του και κάλυψε όλο το φάσμα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η ισότητα αυτή γνώρισε σημαντικές πρόοδους. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλες προσπάθειες στα πλαίσια της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που πλήττει ήδη μια ομάδα του πληθυσμού που ζει ε, σε επισφάλεια, δηλαδή οι γυναίκες. Έχουμε το θέμα θέμα της ε, μειονεξίας του, ότι ανήκουν πολλές φορές σε μια εθνική μειονότητα. Θα ήθελα να επιμένω πάνω σε τρία σημεία. Χρειάζεται να έχουμε δείκτες αξιόπιστους, συνεκτικούς και κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προτείνουμε λύσεις προσαρμοσμένες ε, στην πραγματικότητα με βάση στοιχεία αξιόπιστα σε σχέση με την ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες. Αν θέλουμε πράγματι να έχουμε μια πραγματική ισότητα, θα πρέπει να υπάρχει μια διαπατρότητα ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο επίπεδο. Αυτό είναι σημαντικό για τις ίσες ευκαιρίες στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Η ισότητα περνάει από το γεγονός ότι η γυναίκα πρέπει να ελέγχει το σώμα της. Θα πρέπει να έχει ως το δυνατόν περισσότερη ε, πρόσβαση στην αντισύλληψη και στις αμβλώσεις. Βεβαίως υπάρχουν ε, πάρα πολλέ τριβέ σχετικά με τα θέματα αυτά, αλλά είναι προφανές ότι όσο οι γυναίκες δεν θα μπορούν να ελέγχουν τα σεξουαλικά τους δικαιώματα, δεν θα έχουμε κερδίσει την μάχη για μια πραγματική ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες. Ο Βίρ για ένα λεπτό. Κυρία Οβίρ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφε, θέλω καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Ταραβέλα. Ε, η ο τίτλος ε, «Ισότητα μεταξύ των φύλων» είναι κάτι πολύ γενικό. Στην καθημερινή ζωή πρέπει να υπάρχει ισότητα. Σίγουρα αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με κάποιες μονομένες πράξεις. Εδώ και 40 χρόνια το συζητάμε το θέμα, αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει σημαντική πρόοδος. Το θέμα της εποπτείας και της εφαρμογής των μέτρων είναι επίσης σημαντικό. Ε, παραμένουμε ακόμα σαν γυναίκες σε ένα μεσαιωνικό ρόλο. Θέλουμε να αλλάξει η κατάσταση, θέλουμε να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα. Εμεί αύριο θα εκλέξουμε μια νέα επιτροπή, αλλά μόνο ένα τρίτο των επιτρόπων είναι οι γυναίκες. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε εμείς από σήμερα μέχρι αύριο αλλά θα ήθελα να ζητήσω την επόμενη φορά που θα εκλέξουμε μια επιτροπή να ζητήσουμε όλα τα κράτη-μέλη να υποβάλουν δύο υποψηφίους, έναν άντρα και μια γυναίκα. Και μετά από εκεί και πέρα η απόφαση να ληφθεί βάσει των ικανοτήτων τους και των προσόντων τους. Ε, τα επίπεδα παιδείας αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε κάτι τέτοιο. Και τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σπύρλα για την εργασία του και να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία για το μέλλον. Ευχαριστώ κύριο Στρεμόπουλος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε πολύ σωστά η σημαντική αυτή έκθεση του 2009 αντιλαμβάνεται ότι η βία είναι ένα θεμελιώδες εμπόδιο για την ισότητα γυναικών και ανδρών. Δεν αναφέρεται όμως συγκεκριμένα στην ενδοοικογενειακή βία. Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό βρίσκεται σε έξαρση και μαστίζει όλες τις κοινωνίες. Στην Ελλάδα για παράδειγμα έχουν καταγραφεί μέσα σε 1,5 χρόνο 35 συζυγοκτονίες. Παρ' όλα αυτά οι δομές στήριξης κακοποιημένων γυναικών είναι υποτυπώδεις αν όχι ανύπαρκτες. το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο οφείλει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη φυσικά και την ελλάδα ώστε να δημιουργήσουν δομές στήριξης κακοποιημένων γυναικών σε κάθε δήμο με πλήρη ψυχολογική νομική και επαγγελματική υποστήριξη καθώς και επαρκώς στελεχωμένους ξενώνες για τις γυναίκες επίσης να λάβουν υπόψη τις προτάσεις για τροποποιήσεις που έχουν γίνει από γυναικείες οργανώσεις και νομικούς για νομοθετικές ασάφειες και ελλείψεις γύρω από το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και τέλος να εισαγάγουν προγράμματα αντισεξιστικής εκπαίδευσης στα σχολεία με στόχο την αλλαγή των κοινωνικών αναπαραστάσεων εκείνων δηλαδή ε, που σχετίζονται με τους στερεότυπους κοινωνικούς ρόλους. ευχαριστώ. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριος Πάσκα. Νομίζω ότι ε, η έκθεση είναι σωστή, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με την ισότητα των ανδρών και γυναικών. Αλλά ε, δεν μπορώ να μην πω ότι είναι σχιζοφρενική η κατάσταση. Η Μεντίνα Μάμι 16 ε, χρονών από την Αντιαμάν ε, την ε, Τουρκία θαύτηκε ζωντανή δίπλα στο σπίτι της. Την βρήκανε δύο μέτρα κάτω από την γη στην αυτοψία ε, είδαν ότι υπήρχε ε, χώμα στο, ε, στο πνεύμονες και στο στομάχι της κόρας. Ο πατέρας ομολόγησε ότι μεταξύ των φίλων της υπήρχαν και αγόρια, όχι μόνο κορίτσια και γι' αυτό την έθαψε ζωντανή. Έτσι σκοτώνονται, δολοφονούνται οι γυναίκες με τον τρόπο αυτό αν πάρουμε στα σοβαρά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, πώς μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μια χώρα που έχει τέτοια προσέγγιση ε, προς ε, τις γυναίκες μπορεί να γίνει μέλος της Ευρώπης. Ε, δεν είναι μόνο οι διαφορές ως προς τις αμοιβέ και τους αμυνιστούς. Πρέπει να ασχοληθούμε με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια που δεν ισχύει για τις γυναίκες σε πάρα πολλές χώρες. Ευχαριστώ για ένα λεπτό η κυρία Στάσεν. Σήμερα συζητούμε για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήδη Έχουμε ήδη πει πολλά πράγματα, αλλά αν λείπει ένα στοιχείο είναι η ανισότητα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών ε, στην κοινότητα την ευρωπαϊκή όπου η γυναίκα είναι, ε, υπάγεται στην, ε, στο Ισλάμ, στον άνδρα, στην Ισλαμική κοινότητα την ευρωπαϊκή. Η γυναίκα υπάγεται στον άνδρα, ο Ε, δεν πρέπει η ευρωπαϊκή κοινότητα ε, να καταπολεμάει το δικαίωμα να φοράει κανείς μπουρκα, αλλά το, δικαίωμα να μην φοράει μπουρκα. Ε, στην Γαλλία ψηφίζονται νόμοι, θα ήθελα και εδώ να υπάρξουν οι ίδιοι κανόνες. Δράστε υπέρ των γυναικών αυτών, των μουσουλμανικών γυναικών. Καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις, θα πρέπει να μπορούν να σπουδάσουν ελεύθερα, να μην υπάγονται στους άνδρες, να είναι ελεύθερες να χειραφετηθούν. Θα πρέπει να δράσουμε υπέρ των γυναικών αυτών και είναι ένα στοιχείο που λείπει από την έκθεση του εισηγητή. Ευχαριστώ. Δίνω με τον λόγο στον συνάδελφο Κλάς δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κλάς, ε, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι, για πολλωστή φορά σήμερα σημειώνω ότι οι γυναίκε εξακολουθούν να μην είναι ισότιμε στην Ευρώπη όσον αφορά την εργασία του. 51% ε, το ποσοστό της εργασίας αυξήθηκε σε 58% σήμερα. Είναι πολύ ικανές, έχουν πάρα πολλά προσόντα οι γυναίκες, αλλά δεν έχει αυξηθεί το ποσοστό τους όσον αφορά θέσει, τις ηγετικές θέσεις και ακριβώς όσον αφορά οικονομία νομικά ε, και άλλες παρόμοιες σπουδές το ποσοστό των γυναικών είναι πολύ ψηλότερο. Παρ' αυτό το 2007 το 30% των γυναικών ήταν απασχολούμενες σε μερική απασχόληση, τετραπλάσια αριθμός από ότι οι άντρες και εισπράττουν το 17% λιγότερο από τους άντρες και απειλούν περισσότερο με φτώχεια. Ιδίω μετά τη σύνταξη. Θα πρέπει να αλλάξει η γυναίκη στην οικονομία, η γυναίκη στην εργασία. Ζητούμε ιδιαίτερε ε, ειδικέ θέσεις για να μπορούμε να εξισώσουμε το χρόνο μητρότητα. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι γυναίκε είναι πάρα πολύ ακριβέ και γι' αυτό δεν προσλαμβάνονται. Αυτό οφείλεται όμως στο γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεται πάρα πολύ η εργασία στην οικογένεια. Είπατε θέλετε να ελέγξετε την, ε, το κόστος ε, και όφελος της διαδικασίας αυτής. Αλλά δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε έτσι κύριε Επίτροπε. Ε, γιατί δεν δεχόμαστε ότι κατά βάση θα, οι άνδρες και οι γυναίκες ασχολούν ευχαρίστως με τα παιδιά τους εάν αυτό δεν οδηγεί σε μία μείωση των ε, προοπτικών σταδιοδρομίας. Η οικονομία θα πρέπει να δεσμευτεί υπέρ της οικογένειας, υπέρ των γυναικών. Χρειαζόμαστε μια μετατροπή του σκέφτεστε στην οικονομία, όχι περισσότερους νόμους και θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει κύριε Παδοπούλου για λεπτό. Πρόεδρε, η διεθνή οικονομική κρίση έχει σαφεί αρνητικέ επιπτώσει για άντρε και γυναίκε. Συνεπάγεται απώλεια θέσεων εργασία, επιβάλλει δημοσιονομικέ πολιτικέ λιτότητα σε καμία όμω περίπτωση δεν πρέπει να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στην περαιτέρω προώθηση πολιτικών για την ισότητα ανδρών γυναικών γιατί αυτέ οι πολιτικέ μπορούν να αποτελέσουν την ατμομηχανή για κοινωνικο οικονομική ανάπτυξη και ανάκαμψη στην ευρώπη η κρίση συνιστά παράλληλα μια μοναδική ευκαιρία και πρόκληση για να δημιουργήσει η ευρωπαϊκή ένωση και οι κυβερνήσει των χωρών μελών τη συνθήκε αύξηση τη ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο αναθεωρώντα και ενσωματώνοντα τη διάσταση τη ισότητα των φύλων σε όλε τι πολιτικέ ώστε να αντιμετωπιστούν πάγια δημοκρατικά ελλείμματα σε βάρο τη γυναίκα οφείλουμε να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες για να πατάξουμε την ανισομιστία, τη βία το φαινόμενο της γυάλινης οροφής τις διακρίσεις τη φτώχεια. οφείλουμε να βρούμε τρόπους συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής βελτίωσης των υποδομών φροντίδας παιδιών βρεφών και ηλικιωμένων στήριξης εργαζομένων γυναικών και ζευγαριών διπλής σταδιοδρομίας μονογονιών και ατόμων με αναπηρία πρωτίστως οφείλουμε να θέσουμε σε εφαρμογή με αποτελεσματικότητα όλες τις νομοθεσίες περί στην πράξη. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Χίρς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, με το ευρωπαϊκό Έτο τη Φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού οι γυναίκε έχουν περισσότερε πιθανότητε να είναι φτωχέ και να ζουν σε φτώχεια. Χρειάζονται πολλά μικρά ε, βήματα να βελτιωθούν, γιατί πολλέ φορέ οι γυναίκε επιλέγουν μια θέση εργασία που δεν είναι τόσο αποδοτική ή η απόφαση υπέρ ενός παιδιού που οδηγεί σε μερική απασχόληση ή η απόφαση να φροντίσει κανένα στους γονείς τους, τους παππούδες του πάλι οι γυναίκες δεν έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και να ε, κερδίσουν τη ζωή τους. Όλα αυτά αρθρίζονται και το αποτέλεσμα είναι η επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών να προχωράει με πολύ πολύ μικρά βηματάκια. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και στο μέλλον τους γιατί οι συντάξεις είναι πάρα πολύ χαμηλές. Υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές και στην έκθεση. Αυτό που είναι σημαντικό νομίζω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες πάρα πολλές νομοθετικές δυνατότητες, αλλά θα πρέπει να σε εκμεταλλευτούν οι κοπέλες, οι γυναίκες. Η τόλμη μια κοπέλα να σπουδάσει μηχανολόγος, μηχανικός, αυτό είναι σημαντικό. Και θα ήθελα να τονίσω, όταν δει εδώ κανένα γύρω, έχουμε δύο τρίτα γυναικών, ένα τρίτο ανδρών. Θα πρέπει και οι άντρες να ασχοληθούν με το θέμα αυτό, να προσπίσουν αυτά τα συμφέροντα και να έχουμε περισσότερους άντρες εδώ που να προσπαθούν να βοηθήσουν τις γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Σκριμπλέσκα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, στην έκθεση του κύριου Ταραμπέλα βρίσκουμε έναν αριθμό σημαντικών διατάξεων και παρατηρήσεων σε σχέση με την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Ως προς την ανισότητα βλέπουμε τη διαφορά στους μισθούς και θα πρέπει η διαφορά αυτή να γεφυρωθεί. Οι άντρες που εργάζονται σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις ε, και ε, όπου εργάζονται και γυναίκες που δεν καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση. Έχουμε επίσης ε, και την περίοδο εργασίας που απαιτείται για συνταξιοδότηση. Υπάρχει βεβαίως προσπάθεια να ενταχθούν καλύτερα οι γυναίκες στην αγορά εργασίας όταν θέλουν να επενενταχθούν αφού έχουν αναθρέψει τα παιδιά τους. Θα πρέπει οι επιχειρηματίες να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα αυτό Η έκθεση επίσης δείχνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες, των γυναικών που φροντίζουν άλλα άτομα. Αλλά μεταξύ των θέμων αυτών έχουμε πλεονάζουσες δηλώσεις σχετικά με την αναπαραγωγή και με την, στην, όσον αφορά την ε, την πρόσβαση σε αμβλώσεις χωρίς όρια. Θα πρέπει οι αμβλώσεις να παραμείνουν στην αρμοδιότητα και ευθύνη των κρατών μελών. Η ίση ανδρών και γυναικών δεν πρέπει ε, να συγχέεται με αποφάσεις σχετικά με την σεξουαλική ζωή. Και ε, λόγω των, των θεμάτων αυτών μειώνεται η υποστήριξη αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Μπλίνκεβιτσούτε. Ευχαριστώ τον κύριο Ταραμπέλα για την εργασία που έκανε σχετικά με την οικονομική κρίση ε, θα πρέπει να ενισχυθεί η ανθρώπινη δομή για τις γυναίκες, να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται κοντά στον στόχο της στρατηγικής της Λισαβόνας μέχρι το 2010 το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών. Αλλά από τη μια χώρα στην άλλη η κατάσταση είναι άνηση σχετικά με το θέμα αυτό. Για το λόγο αυτό τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν πρέπει να λάβουν μέτρα ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στον τομέα της εργασίας να, να εφαρμοστεί καλά. Υπάρχουν διαφορές σε ορισμένες χώρες ανάμεσα στους μισθούς ανδρών και γυναικών. Θα πρέπει να κληθούν ε, τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την αρχή για ίση εργασία, ίση αμοιβή. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει νομοθεσία ευρωπαϊκή για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να γίνει καλύτερη κατανομή των καθηκόντων των οικογενειακών και επαγγελματικών, να είναι καλύτερη κατανομή του χρόνου ανάμεσα στην αμοιβόμενη και μη αμοιβόμενη εργασία. Θα πρέπει να υπάρχουν βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί κατάλληλοι. Η άδεια πατρότητας δεν έχει διευθετηθεί. Γι' αυτό πρέπει να βρεθεί μια λύση το συντομότερο δυνατόν να υπάρξει μια οδηγία ως προς το θέμα αυτό σε σχέση με τη νέα στρατηγική για 2020 η διάσταση ανδρών γυναικών είναι απούσα από τη στρατηγική αυτή ενώ θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τον ενεργό του ρόλο στον τομέα που συζητούμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Καλή συνέχεια. Η κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα για δύο λεπτά. Ευρώπη, zachodzą zmiany, jak wynika z raportu, które ε, γίνονται πολλές αλλαγές στην Ευρώπη και αυτό αναφέρει και η έκθεση. Τονίζεται η μετατροπή βασισοποίησης ε, οι γυναίκες έχουν περισσότερη απασχόληση. Αυτό γίνεται ιδίως εκείνες στις οικονομίες όπου οι γυναίκες μπορούν να πάρουν αποφάσεις από πάνω τους, αλλά εκεί που δεν έχουν επίδραση στην εργασία τους, δυστυχώς τα στερεότυπα που επικρατούν δεν τους δίνουν δυνατότητα να δράσουν στην δημόσια ζωή. Γι' αυτό η συμβολή του στην ε, πολιτική είναι πάρα πολύ μικρή. Το πρόβλημα είναι τα στερεότυπα και το Γι' αυτό θα πρέπει να τονίσουμε την ισότητα ανδρών και γυναικών. Η έκθεση τονίζει την ανάγκη να ενδυναμωθούν αυτές οι δράσεις και οι δραστηριότητες. Ακόμα όμως δεν έχουν γίνει αρκετά. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να εξετάσουν το θέμα τη συμβολή των γυναικών στην πολιτική εκεί που οι γυναίκες συμβάλλουν στην πολιτική μπορεί να πετύχουν πολύ καλύτερα την ισότητα ε, ανδρών και γυναικών. Στην Πολωνία αρχίσαμε την συζήτηση όσον αφορά τις ε, προτεραιότητες και τις πολιτικές και υπήρχε μια ομάδα γυναικών που συζήτησε το θέμα και θα θέλουμε αυτό να προχωρήσει. Θέλαμε το 50% των γυναικών να είναι στις εκλογικές λίστες, μάλλον οι εκλογικές λίστες να αποτελούν κατά 50% από γυναίκες. Συζητούμε το θέμα αυτό και χωρίς να μπορούμε να ε, γνωρίζουμε κατά πόσο τελικά η Πολωνική Βουλή θα υπερψηφίσει, θα καταψηφίσει οι παρόμοιες προτάσεις, Όλο αυτό το θέμα της συζήτησης είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό θα ήθελα να σας πω ότι θα ήταν καλό να συζητήσουμε το θέμα της συμβολής των γυναικών στην πολιτική στην Ευρώπη. Πρώτα, ευχαριστώ. είναι εσύ για ένα λεπτό. Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε το θέμα του ότι οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν τον έλεγχο της σεξουαλικής ζωής τους, της αναπαραγωγής και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην αντισύλληψη και σε μια ασφαλή άμβλωση. Στην Πολωνία το δικαίωμα το πολιτικά δικαιώματα έχουν σχέση, επηρεάζουν ε, την αντισύλληψη και την άμβλωση. Ε, δεν μιλούμε για άμβλωση, αλλά μιλούμε για δολοφονία ενός παιδιού που έχει συλληφθεί. Και υπάρχουν προσπάθειες να η πρόληψη της άμβλωσης να περιληφθεί στο Σύνταγμα. Οι άνθρωποι έχουν ειδοποιηθεί ότι δεν υπάρχει θέμα αμβλώσεων. Ε, υπάρχει Ευχαριστώ, το δικαίωμα αναπαραγωγή ε, των γυναικών. Κύριε Χύπνερ, δύο λεπτά. Η κυρία Χύπνερ έχει το λόγο. Ε, Frau Kollegin Hübner hat das Wort für zwei Minuten. Η συνάδελφος Χίμπνερ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Uh, represent half of Οι γυναίκε προσωπούν το 5% του ε, ταλέντου στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να τις παραβλέψουμε γιατί εάν τις εκμεταλλευτούμε στην οικονομία θα κάνουμε ένα τεράστιο άλμα προς τα και όσον αφορά την ενεμετώπιση στην ε, Ευρώπη όσον αφορά τις νοοτροπίες και όσον αφορά τις δυνατότητες. Η ισότητα των ευκαιρών υπάρχει επί χάρτου τουλάχιστον. 13 οδηγίες έχει προετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. Στην πραγματικότητα όμως η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Ποτέ δεν ήταν τόσο καλά εκπαιδευμένες οι γυναίκες, αλλά όσον αφορά τις επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην εκπροσωπούν σωστό. Υπάρχει ένα κενό φύλλο αυτή τη στιγμή. Οι γυναίκες, ε, αν δανειστούν χρήματα, τα επιστρέφουν οπωσδήποτε. Παρόλα αυτά έχουν δυσκολίες να έχουν πρόσβαση σε χρήματα. Χρειάζονται περισσότερα χρήματα να μπορούν να δανειστούν χρήματα. Αλλά μόνο το 1% των περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο είναι στα χέρια γυναικών οι γυναίκες εξακολουθούν να μην εκπροσωπούν σωστά όσον αφορά εκείνους που λαμβάνουν αποφάσεις. Θα πρέπει οι γυναίκες να παίξουν εκεί ένα ρόλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μόνο έτσι οι γυναίκες θα μπορέσουμε να προχωρήσουν. Η πραγματική ισχύ βρίσκεται στο θέμα της λήψης αποφάσεων. Θα πρέπει πολλά να γίνουν για να αλλάξουν. Μία γυναίκα σε ένα σώμα λήψη απόφαση θα πρέπει να αλλάξει η στάση τη για να προσαρμοστεί στην πλειοψηφία των εδρών. Πολλέ γυναίκε σε τέτοιε θέσει θα ε, οδηγούσαν σε κάποιε αλλαγέ. Θα πρέπει όμω να άρουμε το μεγαλύτερο εμπόδιο τη γυναίκα, δηλαδή η συμφιλίωση τη επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Χρειαζόμαστε πολιτικέ, οι οποίε προσανατολίζονται στο θέμα του φύλου και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η Ζάφος Παλεντέλ έχει το λόγο. Frau Kollegin Paledelli ist nicht da, dann kommt als nächstes. Απουσιάζει κυρία Παλεντέλη. Η κυρία Παπα-Νικολάου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ενώνω και εγώ σήμερα τη φωνή μου με τη φωνή των συναδέλφων, των πολλών γυναικών και των όχι όμως και τόσο λίγων ανδρών και με τον άντρα εισηγητή μα, τον κύριο Ταραμπέλα τον οποίο συγχαίρω και δηλώνω και εγώ ότι όλοι μας στηρίζουμε με πάθος κάθε δράση, κάθε πρωτοβουλία για την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και αυτό είναι αυτονόητο γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούμε σε μια ανοιχτή δημοκρατική φιλελεύθερη κοινωνία στην οποία καθένας από εμά θέλει να ζει. γίνεται σημαντική προσπάθεια και αυτό πρέπει να το τονίζουμε. σε ευρωπαϊκό επίπεδο θυμίζω την οδηγία 54 του 2006 που όριζε την εξάλληψη κάθε μορφής διάκρισης μεταξύ των δύο φύλων από τα κράτη μέλη μέχρι τον αύγουστο του 2009 θυμίζω επίσης τον ευρωπαϊκό χάρτη Αξιολόγησης που εξέδωσε η επιτροπή για την καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων εντό ευρωπαϊκή ένωση από την περίοδο του 2006 μέχρι το. 2010. θυμίζω επίσης και θέλω να συγχαρώ γι' αυτό κάθε πρωτοβουλία εθνικών κυβερνήσεων στα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης με τελευταία αυτήν της γαλλικής κυβέρνησης και του προέδρου σαρκοζή σε σχέση με την προώθηση νομοθεσίας για την απαγόρευση της μπουρκας στους δημόσιους χώρους όλα αυτά είναι βήματα χρειάζονται όμως ακόμη περισσότερα προκειμένου να αλλάξουμε πάνω απ' όλα την οτροπία μας σε σχέση με την αποφυγή κάθε διάκρισης που παρατηρείται και δυστυχώς υπάρχουν ακόμη διακρίσεις και επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά σε μια ευαίσθητη κατηγορία σε αυτή των νέων μητέρων διαβάζω με έκπληξη σε έκθεση της ευρωπαϊκής επιτροπής σε σχέση με τους στόχους της βαρκελώνης για την φροντίδα των παιδιών στην ευρωπαϊκή ένωση ότι σχεδόν το σύνολο των ευρωπαίων μητέρων δηλώνουν αδυναμία να αναθρέψουν όπως επιθυμούν τα παιδιά τους εξαιτίας των υπέρογκων ευθυνών που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε και εδώ να δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή έμφαση ότι η αδυναμία επίτευξης πραγματικής ισότητας μεταξύ των δύο φύλων θέτει σε κίνδυνο τα σημερινά παιδιά που στερούνται ένα ισορροπημένο οικογενειακό περιβάλλον με έντονη τη μητρική παρουσία. θέτει σε κίνδυνο την ψυχική ισορροπία και την ανάπτυξη συγκροτημένης προσωπικότητας των σημερινών παιδιών και των αυριανών πολιτών της ευρωπαϊκής ένωσης. σας ευχαριστώ πολύ. Γκούρμα το λόγο. Η οικονομική κρίση ε, κατέδειξε ότι τα θέματα της οικονομικής ανεξαρτησίας είναι πολύ στενά συνδεδεμένα με τα θέματα της ισότητας. Αυτό το είδαμε ανάλογα με το πώς έχουν πληγεί ορισμένες χώρες από την κρίση αυτή ρόλο τη γυναίκα ε, στην οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει όμω να λάβει η Κομισιόν ε, μια πολύ αυστηρή θέση όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων και να προσανατολίσει όλε τι πολιτικέ εκεί. Όπω ο Σάνφος Ταραμπόλα τόνισε στην έκθεσή του, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να προωθήσουμε την οικονομική και κοινωνική θέση των γυναικών. Θα πρέπει να δώσουμε να δώσουμε κάθε δυνατότητα συνέντες. Τελευταία ευκαιρία να σας πούμε γεια σας κύριε Σπίτλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή σας. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ συνάδελφο Πάνω και δύο λεπτά. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι... όλα ελέγχθησαν σε αυτή τη τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω εγώ να παρουσιάσω μια νέα πτυχή, κάτι θα μπορούσα ίσως να παρατηρήσω. Θα πρέπει για όλους μας εμάς να είναι στόχος οι γυναίκες να μην ε, αναγκάζονται να επιλέξουν άμεσα σε οικογένεια και σε επάγγελμα. Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσουν να συμφιλειώσουν τα δύο αυτά. Θα πρέπει στο μέλλον να υιοθετηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε το σώσει μια γυναίκα να μπορεί να παίξει το ρόλο της αφενός ως μητέρα και αφετέρου στην δουλειά της, ε, στην οικονομία. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σχήμα μισοδότησης ισότιμο. Θα πρέπει ο χρόνος που χάνουν με την ανατροφή των παιδιών να μπορεί να ε, καλύπτεται αργότερα. Νομίζω ότι αυτή η λύση είναι μια λύση που θα πρέπει να έχουμε κατά νου, ιδίως σε οικονομικά δύσκολους καιρούς. Και αν καταφέρουμε και μπορούμε εμείς ως Κοινοβούλιο πολλά να συμβάλλουμε, θα πετύχουμε μία σύγχρονη και ισότιμη Ευρώπη. Γιατί αυτό είναι δυνατό μόνο με την ισοτιμία ανδρών και γυναικών. Ευχαριστώ. Πρώτα σε ευχαριστώ συνάδελφε. Η συνάδελφος Τόμψεν, 1,5 λεπτό. Η έκθεση Ταραμπέλα για την ισότητα δείχνει με λαμπρό τρόπο τις τεράστιες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία από αυτές τις προκλήσεις είναι η συμμετοχή των γυναικών στις, ε, στον επιχειρηματικό βίο, στα διοικητικά συμβούλια των ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Σε περίοδο χρήσης πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα ταλέντα. Να πάρουμε το μάθημα από την Νορβηγία όπου η Νορβηγή, ο Νορβηγός Υπουργός Οικονομίας ζήτησε 40% των γυναικών να συμμετέχουν στον οικονομικό τομέα διότι για να αντιμετωπίσουμε την ανταγωνιστικότητα χρειάζεται ισότητα των φύλων. Εμείς ε, λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό από όλα τα φύλλα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη. Παράδειγμα λοιπόν από τους Νορβηγούς. 200 Νορβηγίδες συμμετείχαν ως επικεφαλής επιχειρήσεων ή στελέχη και στις επιχειρήσεις όπου έχουμε ισότητα των φύλων η οικονομική κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από ό,τι αλλού ίση λοιπόν αντιπροσώπευση. Ο κύριος Κασίνη. Ευχαριστώ. Η αρχή ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών εντάσσεται με... μπαίνει μάλλον στο γενικό ρεύμα αυτού του μεγάλου ποταμού που αλευθέρωσε σκλάβους άντρες, γυναίκες, εργάτες κλπ. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική έκθεση τα Ταραμπέλα. Αλλά δύο παρατηρήσεις. Η ανθρώπινη ισότητα πρέπει να αφορά όλους, ακόμη και τα παιδιά που δεν έχουν ακόμη γεννηθεί. Είναι παράδεκτο να λέμε στο σημείο 38 να αγιοποιούμε την άμβλωση θεωρώντας τις απαράβατο σεξουαλικό δικαίωμα των γυναικών. Εντάξει, κανένας δεν αρνείται τα προβλήματα των δύσκολων εγκυμοσυνών <coughs> των ε, προβλημάτων υγείας. Πρέπει όμως να δίνουμε τη δυνατότητα της, της ελεύθερης επιλογής στις γυναίκες. Και επίσης θα πρέπει να αναφερόμαστε και στις κοινωνικές πτυχές της εγκυμοσύνης. Τι σημαίνει οποιαδήποτε σεξουαλική συμπεριφορά, όποια και να είναι, θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να επενείται κάθε φορά όπως και να έχει. Μα έτσι δεν φύγουμε και το θέμα της ελεύθερης γνώμης και της ελεύθερης συνείδησης. Αυτά είναι τα ερωτηματικά μου που νομίζω ότι δεν είναι μπανάλ. Λοιπόν, catch the eye. Η κυρία Μαγκίνες για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλοί λένε ότι η περισσότερη νομοθεσία δεν είναι η λύση αν δεν εφαρμόσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία. Επίσης, η κίνηση για περισσότερη ισότητα πολύ συχνά οι γυναίκες θεωρούν ότι η μάχη έχει τελειώσει. Θα πρέπει να εμψυχώσουμε τους νέους και τις νέες για την οικονομική κρίση βεβαίως επηρεάζει τις ε, γυναίκες. Αλλά όταν ο άνδρας χάνει τη δουλειά του επίσης επηρεάζεται η γυναίκα. Η οικονομική κρίση πλήττει όλους, κυρίως τις οικογένειες. Στις παράγραφους 34 και 35 συμφωνώ πλήρως και θα πρέπει ε, να επικυρώσουμε τις ε, συμβάσεις ε, που υπάρχουν οι χώρες που δεν τις έχουν επικυρώσει. Σχετικά με την οικογενειακή βία και πάρα πολλές γυναίκες δολοφονούνται μέσα στο σπίτι τους Είχαμε και στην Ιρλανδία μια τέτοια περίπτωση στα δικαστήρια. Για την παράγραφο 38 βεβαίως θα πρέπει σε σχέση με τις αμβλώσεις να σεμβαστούμε την επικουρικότητα και χρειάζεται η παράγραφος αυτή τροπολογία. Η κυρία Σινάλοβα για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ και 100 χρόνια περίπου οι γυναίκες ήθελαν ε, τα δικαιώματά τους ε, να γίνουν σεβαστά. Αυτό ισχύει και σήμερα νομίζω. Κυρίως ε, να πρέπει οι γυναίκες να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή και να έχουν ίσες συνθήκες ακόμα και στην πολιτική ζωή. Νομίζω ότι στις τελευταίες εκλογές στην Τσεχική Δημοκρατία ο ρυθμός των γυναικών αυξήθηκε από 15% σε 26% και μπορούμε να έχουμε παρόμοια παραδείγματα στις άλλες χώρες. Οι ε, γυναίκες δεν θα ζητήσουν τίποτα αν έχουν ίσα δικαιώματα και θα είναι πάρα πολύ δραστήριες αν έχουν ίσα δικαιώματα. Αν οι γυναίκες δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην πολιτική ζωή, δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε για ίσες ευκαιρίες. Γι' αυτό θα πρέπει να αγωνιστούμε για ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες και τότε δεν θα ε, χρειαστούμε ε, ποσοστώσεις. Κύριε, πριν από μερικά λίγο καιρό έκανα μια ομιλία στη Γερμανία όσον αφορά τις εργασίες μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και το τι κάνω. Και ένα άντρα με ρώτησε και τι λέει ο άντρας σας επ' αυτού. Ξέρω ότι αυτή η ερώτηση υποβάλλεται πολύ συχνά. Σε αντίθετη περίπτωση κανέναν άντρα δεν ρωτάνε. Και η γυναίκα σας τι είπε. Μια άλλη περίπτωση. Ε, ναι, ένα νερό ζευγάρι που απέξε ένα παιδί και τα δύο παιδιά αυτά μοιράζονται μία θέση απασχόλησης για τη γυναίκα αυτό γίνεται, έγινε δεκτό. Ε, ο άντρα ερωτήθηκε, μα γιατί κάθε και αλλάζει πάνε στη μισή μέρα. Και τι σχέση έχει αυτό με την ε, σταδιοδρύμη σου. Μετά εξετάσαμε το θέμα των ε, επιχειρήσεων. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στις οποίες οι γυναίκες δεν έχουν τη δυνατότητα να ξαδιοδρομήσουν. Και τέλος, σε εταιρείες στις οποίες τουλάχιστον 30% ε, είναι στη διαχείριση ε, έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Καταλάβατε ότι η ισότητα ισχύει και όσον αφορά το χρόνο αγόρευσης. Κυρία Νικολέσκου έχει το λόγο. Ο κύριος Νικολέσκου. Αυτή η έκθεση είναι πάρα πολύ καλή, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε το ρόλο της αγρότησας τόσο όσον αφορά την καθημερινή της δουλειά, όσο και την εισφορά της στην οικογενειακή οικονομία. Και είναι μάλιστα και προτεραιότητα η αγρότησα για την Ισπανική Προεδρία. Και θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ρόλος της μέσα στα πλαίσια της Ατζέντας 2020 που θα συζητηθεί στις Βρυξέλλες αυτήν την εβδομάδα. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Κάτεμπακ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τεραβέλα. Νομίζω ότι το ότι είναι πάνω από 40 χρόνια αποδεικνύουν ότι το θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να εξετάσουμε σε, μια ώρα. Είναι ένα θέμα που αξίζει πάρα πολύ συζήτηση. Εγώ θα συγκεντρωθώ σε δύο σημεία. Το σημείο 8 που ε, επικρίνει το θέμα ότι το mainstreaming των ισοτιμίας ε, ε, δεν λαμβάνεται υπόψη στην πολιτική της και θα ήθελα να το λάβει υπόψη της Κομισιόν για τη μελλοντική της πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Επίσης, Νομίζω ότι τα κρατη μελη μπορούν να κάνουν μια αξιολόγηση των επιπτώσεων, γιατί εάν θέλουν να καταπολεμήσουν τις επιπτώσεις της κρίσης, χρειάζονται μέτρα τα οποία λαμβάνουν υπόψη την ειδική κατάσταση των γυναικών. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να κληθούν τα κράτη-μέλη βάσει των στοιχείων αυτών να ε, υιοθετήσουν κάποια μέτρα για την πρόθεση της οικονομικής ανάπτυξης. Θεωρώ ότι οι γυναίκες έχουν επίσης δικαίωμα να ελέγχουν το σώμα τους και την υγεία τους. Ευχαριστώ. Στην Αλφας Νικολά έχει το λόγο. Domnule președinte, apreciind raportul, vreau să subliniez την έκθεση, θα ήθελα να πω το εξή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η νομοθεσία στον τομέα αυτό, γιατί η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι ε, ε, ένας ουσιαστικός ε, παράγοντας του πολιτισμού και της παράδοσης στα κράτη-μέλη και γι' αυτό θα πρέπει να θετηθούν θετικά μέτρα κατά τέτοιο τρόπο ούτω ώστε από πολύ νωρίς να μαθαίνουν τα παιδιά τι γίνεται και να αποφεύγουν τη στερεότυπα μια κουλτούρα ισότητας ανδρών και γυναικών θα πρέπει να ε, υπάρχει από την πιο μικρή ηλικία. Αλλιώς δεν θα πετύχουμε και θα έχουμε και στο μέλλον τις ίδιες συζητήσεις. Και το μόνο που θα μπορούμε να δούμε στο μέλλον είναι ότι υπάρχει ανισότης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σε ένα πολιτισμό γνώσης, σε μια νέα η οικονομία θα πρέπει να αποφευχθούν αυτές οι διακρίσεις. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Λέτοβα. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι οι στόχοι της Βαρκελόνης δεν ε, ε, συμφωνούν με τα όσα λένε οι εμπειρογνώμονες. Ε, Πιστεύουν ότι οι εμπειρογνώμονες, ότι τα μικρά παιδιά ε, μέχρι δύο ετών δεν θα πρέπει να τη χάνουν φροντίδας εξωτερικής διότι θα πρέπει ο πατέρας ή η μητέρας να φροντίζουν όλη την ημέρα για αυτά τα πολύ μικρά παιδιά. έχουμε τα δικαιώματα των κρατών μελών και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε μέτρα ευρωπαϊκά αποτελεσματικά για να καταπολεμήσουμε ε, την λαθρέα διακίνηση των ανθρώπων και νομίζω ότι η έκθεση αυτή ε, δεν τιμά τα δικαιώματα των μη γεννημένων, των αγέννητων ακόμα παιδιών και ε, θα ήθελα κατά κλείδι να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Σπίτλα ε, και να του ευχηθώ πολύ επιτυχία στη μελλοντική του εργασία. Ευχαριστώ συνάδελφε την Έλαβα. Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Χρειάστηκαν επί 30 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πολλά για το καθεστώς των γυναικών και τα δικαιώματά τους. Υπάρχουν όμως πολλές διαφορές όσον αφορά την αμοιβή. Υπάρχει ένα χάσμα ως προς την αμοιβή, μια τεράστια διαφορά και αυτό έχει να κάνει ε, με την ζωή των γυναικών και αυτή, αυτή η διαφορά σχετίζεται με, με διαφορετικά ε, κοινωνικά ε, θέματα. Θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή καμπάνια ούτως ώστε να εξαλειφθούν οι παλιές προκαταλήψεις που λένε ότι αυτοί που φοράνε παντελόνια είναι καλύτεροι και αυτοί που φοράνε φούστες και αυτές που φοράνε φούστες είναι χειρότερες. Αυτά τα πράγματα είναι ακόμα ταμπού. Θα πρότεινα επίσης τα θέματα ίσων ευκαιριών θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα προγράμματα των δημοτικών σχολείων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 έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κοινωνικό δυναμικό που δεν το εκμεταλλευόμαστε και θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στο μέλλον για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί η κοινωνία. Οι γυναίκες είναι καλύτερα εκπαιδευμένες, αλλά δεν προωθούνται όσον αφορά παραδείγμα, τις χαριστατικές επιστήμες. Θα πρέπει να τις προωθήσουμε όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην πολιτική. Είναι καλές στην ε, διαχείριση, αλλά η συμμετοχή τους σε μεγάλες επιχειρήσεις είναι μικρές. Θα πρέπει οι γυναίκες επίσης να εμπλακούν περισσότερο στην προώθηση καλών πρακτικών και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Σπίτλαρ που μας δίνει την δυνατότητα Ευρωπαϊκού Ταμείου Επένδυσης στην νηπιαγωγία και εάν έχω ένα παιδί κατά τη διάρκεια της θητείας μου θα είμαι πολύ ευτυχής να μπορέσω να το δώσω στην, ε, στο βρεωτικό σταθμό εδώ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Τίκαο έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πετροπέ. Για, για να έχουμε ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών, χρειάζεται και ίσες δυνατότητες σταδιοδρομίας. Χρειαζόμαστε παιδικούς σταθμούς, διότι εδώ υπάρχει λίστα αναμονής για να γραφτεί κάποιος στον παιδικό σταθμό. Δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί. Χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη δημιουργία των παιδικών σταθμών, να υπάρξει κοινωνική πολιτική σχετικά και να γίνουν σχετικές επενδύσεις. Επίσης, τι γίνεται με τις μονογονικές οικογένειες που δεν έχουν τέτοιου είδους υποδομή. Szanowny panie przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy. Υπάρχουν δύο κλειδιά για την επίδευση της ισότητας ανδρών και γυναικών. Το ένα κλειδί είναι η ίση πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία και η δεύτερη είναι πρόσβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δεν επιτρέπεται να συνεχίσουμε να έχουμε αυτές τις διάφορες ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών για την εργασία τους θα πρέπει οι γυναίκες να πληρώνουν το ίδιο όπως και οι άντρες. Θα πρέπει να τονίσουμε την μεγαλύτερη συμβολή των γυναικών στην οικονομική και πολιτική και κοινωνική ζωή. Και νομίζω ότι εάν περισσότερες γυναίκες συνέβαλαν στην πολιτική ζωή θα είχαμε μια διαφορετική κατάσταση. Και όλα μας τα σχέδια θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα ευθυγρασμένα με τα όνειρα και τις προσδοκίες όλες της κοινωνίας. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Πασέσκου. Σε αυτήν την χρηματοπιστωτική κρίση το πόσο στο ανεργία των γυναικών έχει αυξηθεί κατά 1,6% παραπάνω από ό,τι αυξήθηκε η ανδρική ανεργία. Βέβαια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 31% που ήταν οι γυναίκες ε, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία έχουμε περάσει σήμερα στο 35-36 και η Ρουμανία αντιπροσωπεύεται εδώ με το 30% των γυναικών. Αφήστε δε που μία πρώην Ευρωβουλευτήνα είναι πρόεδρος της Ρουμανικής Βουλής και εγώ ως ανεξάρτητη παρουσιάστηκα και με εξέλεξαν παρόλο που είμαι γυναίκα. Οι γυναίκες λοιπόν θα καλύτερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ό,τι στο παρελθόν. Τώρα θα ακούσουμε δύο άντρε. Στην Άλφα Σκέλη πρώτα. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο θέμα μας είναι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι ομιλητές είπαν ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες. Όπως είπε η κυρία Λούλινγκ, έχουν δοθεί πολλές υποσχέσεις από το 1975. Λέγανε ότι οι γυναίκες έχουν κατώτερο ρόλο. Αυτό ισχύει σε πάρα πολλές χώρες. Ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτύχει πολλές πρόοδους. Υπάρχει μια νομοθεσία με στόχους, με κατεύθυνση. Θα έπρεπε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες ε, στους νέους, στα νέα παιδιά, για τα νέα αγόρια. Έχουμε πολύ κακό που γίνεται από εκπομπές τηλεοπτικές και έχουμε έτσι ε, μια άνηση κοινωνία. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Σισάστηκε για να κλείσουμε το ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Zazwyczaj tak jest, że w trudnych czasach więcej problemów z zapewnieniem codziennego bytu rodzinie spoczywa na kobietach. Za to powinno... Υπό δύσκολου όρου συμβάνουν οι γυναίκε πάρα πολύ στην εργασία. Θα πρέπει να το εκφράσουμε αυτό, να εκφράσουμε την ευγνωμοσία μας ε, και να αναφέρουμε και τις κοινωνικές πολιτικές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Πολλά πρέπει να γίνουν στην κατεύθυνση αυτή. Η δημιουργία νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών ίσως ε, σημαίνει ότι δεν συμφωνούμε με τις αρχές. Πολλά μπορούμε να επιτύχουμε για την ισότητα ανδρών και γυναικών στα πλαίσια της παιδείας. Δεν υπάρχει δυνατότητα να εκφράσουμε με έγγραφα το σεβασμό μας προς τις γυναίκες αν δεν υπάρχει αυτό στην κουλτούρα μας, στην Πολωνία λέμε ότι μια γυναίκα στηρίζει και τις τέσσερις γωνιές του σπιτιού. Δηλαδή οι γυναίκες θεωρούνται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές. Το λόγο έχει ο Σπίτλα. Ε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση ήταν πάρα πολύ πλούσια, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχω γνωρίσει πολλές συζητήσεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά νομίζω ότι αυτή η συζήτηση ήταν από τις πιο πλούσιες. η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι η πολιτική αυτή έχει την δική της σημασία και το δικό της προσανατολισμό που πρέπει να ακολουθήσουμε. Όσον αφορά την ισότητα μεταξύ των φίλων και τις ίσες ευκαιρίες, αυτό είναι το επίκεντρο ε, των δικαιωμάτων που πρέπει να εξασφαλίσουμε. Πρέπει η ισότητα να είναι για όλους και δεν θα υπάρχει, ε, δεν πρέπει να υπάρχουν ε, μικρά, μικρές νησίδες όπου δεν ισχύει η ισότητα μεταξύ των φύλων. Η πολιτική που διατυπώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρόγραμμά μας για την ισότητα των φύλων πρέπει να ακολουθήσει αυτόν τον προσανατολισμό. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020 θα περιλαμβάνει περισσότερα μέτρα για την στρατηγική των ίσων ευκαιριών. Πολλοί ομιλητές ανέφεραν ότι μια σύγχρονη κοινωνία η οποία θέλει να είναι επιτυχημένη πρέπει να χρησιμοποιεί όλες τις ανθρώπινες δυνατότητες που έχει. Η ισότητα των φίλων και οι ίσες ευκαιρίες είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Κυρίες και κύριοι, Μιλάμε επίσης ε, για διάφορα μέτρα, για ε, πολιτιστικές απόψεις, για νομοθεσία και για άλλες απόψεις που σχετίζονται με το θέμα αυτό, με το περιεκτικό αυτό θέμα. Όλα τα μέσα είναι ε, διαθέσιμα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υλοποιήσουμε, να εφαρμόσουμε καλά την ισχύουσα νομοθεσία και δεν θα πρέπει να αφιστούμε καμιά προσπάθεια γι' αυτό. Υπάρχουν ακόμα πολλά που απομένει να γίνουν. Βεβαίως καμιά φορά μια νέα θαραλέα νομοθεσία μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Πολλοί ανέφεραν την, την, την Νορβηγία σχετικά με την εκπροσώπηση των ε, γυναικών στις μεγάλες επιχειρήσεις και αλλού. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναλύσουμε αυτό το νορβηγικό παράδειγμα ως προς την υλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Αυτό είναι ένα μέσο εργαλείο πάρα πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Κυρίες και κύριοι, αυτό που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Αυτό είναι ουσιαστικό. Οι ίσες ευκαιρίες είναι κάτι ε, το οποίο ισχύει εξίσου για τους γυναίκες και τους άνδρες. Γι' αυτό χαίρομαι πολύ, πράγματι χαίρομαι πολύ που όλοι συμμετείχαμε σε αυτή τη συζήτηση και όλοι συμβάλαμε και τα δύο φύλλα και οι άνδρες και οι γυναίκες σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό είναι σημαντικό για όλες τις συζητήσεις κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για αυτήν την ευκαιρία που μου δώσατε να βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι η τελική επίσημη παρουσία μου εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Σπίτλα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ όπως και άλλοι συνάδελφοι και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στο μέλλον. Τελευταία θα ακούσουμε τώρα για μια φορά τον εισηγητή, τον κύριο Ταραμπέλα. Και εγώ να ευχαριστήσω για αυτή την τελευταία του παρουσίαση τον ε, Επίτροπο, τον οποίο συνάντησα και άλλες φορές αλλού. Ευχαριστώ όλους για αυτόν τον πλούσιο διάλογο. Τοποθετήθηκαν ένα σωρό συνάδελφοι, τους άκουσα όλους πολύ προσεκτικά. Και χάρηκα που μίλησαν και ένα σωρό γυναίκες, ε, συγγνώμη άντρες. Στην Επιτροπή Γυναικών είμαστε τέσσερις μόνο και οι υπόλοιποι στους 61 είναι γυναίκες. Χάρηκα πολύ λοιπόν που άκουσα άντρες να μιλάνε εδώ μέσα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους. Η κυρία Λούλινγκ έλεγε ότι δεν ήταν άνετη η πλειοψηφία. Στην Επιτροπή 15-8 και 7 αποχές δεν νομίζω ότι ήταν άνισο. Τώρα, για το 38 σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, αντισύλληψη και έκτρωση. Εγώ ξέρω ότι είναι ένα θέμα πολύ πιο λεπτό από ό,τι τα άλλα εγώ δεν μπορούσα όμως ε, να το αγνοήσω το θέμα, έστω και αν δεν ήθελα να βάλω τα πάντα μέσα και αναφέρομαι ε, εδώ στο, στα προβλήματα των ε, κοριτσιών, εφήβων που δεν ξέρουν πώς να τα αντιμετωπίσουν το θέμα και είναι υποκρισία το να, γνωρούμε, να αυτά τα προβλήματα των νέων εφήβων γιατί ε, όταν ε, στους πιο πλούσιους άμα συμβεί κάτι τέτοιο το να ε, δίνεται δυνατότητα στα παιδιά τους για μια αναζωογονητική κούρα στην Ελβετία είναι κάτι το πολύ υποκριτικό. Έχω μερικά δευτερόλεπτα, λοιπόν ξέρετε ότι είναι ένα ντοσιέ το οποίο δεν, στο οποίο δεν μπορούμε να τα χώσουμε όλα. Μιλήσαμε για τις μπουρκες, για τους υποχρεωτικούς γάμους, για όλα αυτά. Λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά ότι στη δημοκρατία ε, αυτού του είδους οι πρακτικές σίγουρα δεν είναι, δεν είναι σεβαστές. Αλλά πιστεύω ότι αν τα είχα βάλει όλα στην έκθεσή μου θα αποπροσανατολιζότανε. Ευχαριστώ κύριε Ταραμπέλα. Ολοκληρώνω τη συζήτηση εδώ. Η ψηφοφορία θα γίνει την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, όχι αύριο. Η επόμενη συνεδρία είναι αύριο, 3η 9 Φεβρουαρίου, 9 με 12.30, 13 και 30, 15 και 30 και 15 έως 20.